Thank Συνάδελφοι, ο κύριος Έλμερ ζήτησε το λόγο για διαδικαστικό. Κύριε Πρόεδρε, η πρώτη παρέμβαση που έγινε ποτέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από εκλεγμένο Ευρωβουλευτή ήταν από τον ε, επίσκοπο Dr. Impaisley το 1979 που επέστησε το γεγονός ότι η Βρετανική σημαία ε, ήταν κρεβεσμένη ανάποδα